Liebe Kolleginnen und Kollegen, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καλωσορίσω ενθέρμως τον υποψήφιο υπο... Επίτροπο για τα θέματα μεταφορών, τον κύριο Μάρο Σέσκοβιτς. Και θέλω να σας ότι ο στόχος της σημερινής ε, ακρόασης βάσει του κανονισμού μας είναι να δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να κρίνει τον ε, υποψήφιο από τη βάση της ικανότητάς του, της δέσμευσή του σε σχέση με την ευρωπαϊκή ιδέα και της ανεξαρτησίας του. Φυσικά θα πρέπει να εξετάσουμε και τις γνώσεις του στον τομέα του επιστητού που θα αναλάβει και την ικανότητα επικοινωνίας του. Θέλω περαιτέρω να αναφέρω ότι στην ε, ακρόασή μας θα λάβουν μέρος και βουλευτές από την Επιτροπή Ήτρα για να θέσουν ερωτήματα σε σχέση με τη διαστημική πολιτική. Η Ήτρε λοιπόν συμμετέχει σε αυτή την ακρόαση. Επίσης θέλω να σας πεθυμίσω ότι ο κύριος Σεύκοβιτς έχει δώσει γραπτές απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσαμε και οι ερωτήσεις αυτές και οι καθώς και απαντήσεις έχουν διανοηθεί στους βουλευτές. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Προτού λοιπόν δώσω το λόγο στον υποψήφιο κύριο Επίτροπο, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να κάνω κάποιε διαδικαστικού χαρακτήρα παρατηρήσει. Η ακρόασή μα θα ακολουθήσει την μέθοδο ping-pong. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ερώτηση θα ακολουθηθεί από μία απάντηση. Θα έχουμε δύο γύρους ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο πρώτος αφορά τους συντονιστές, με συνολικό χρόνο 5 λεπτά για κάθε ερώτηση. Για όλους τους άλλους βουλευτές ο χρόνος θα είναι 3 λεπτά. Και να λάβετε υπόψη σας ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ στενός. Επομένως, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι θα εμφανίζεται ο χρόνος, η αντίστοφη μέτρηση στις οθόνες. Εγώ θα διακόψω όποιον ξεπερνάει το χρόνο και αυτό ισχύει και για τον υποψήφιο κύριο Επίτροπο. Παρακαλώ να τηρήσετε λοιπόν το χρόνο ομιλία σας. Στον πρώτο γύρο θα έχουν οι συντονιστές 5 λεπτά σύνολο. Μπορούν να θέσουν μια ερώτηση το πολύ 2 λεπτών και ο αρμόδιος, ο υποψήφιος επίτροπος θα πρέπει να απαντήσει. Έχει χρόνο να απαντήσει τρία λεπτά το maximum. Να έχετε λοιπόν αυτό υπόψη σας, ότι όσο μακρότερη είναι η ερώτησή σας, τόσο πιο σύντομη θα είναι η απάντηση του Επιτρόπου. Εν τη συντομία η αρετή. Εάν λοιπόν δεν, υπάρχει, δεν έχει εξαντληθεί ο χρόνος των πέντε λεπτών, θα υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής ερώτησης. Αλλά οι συμπληρωματικέ ερωτήσει δεν μπορούν να διεξέλθουν άλλο θέμα από αυτό τη αρχική ερώτηση. Δεν μπορούν να εισαγάγουν ένα νέο θέμα. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ ω πρόεδρο θα είμαι υποχρεωμένο να διακόψω και να αναλάβω να αφαιρέσω το λόγο από τον αρμόδιο συντονιστή. Στο δεύτερο γύρο θα έχουν οι βουλευτές τρία λεπτά για ερώτηση και απάντηση. Και εδώ θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι όσο πιο σύντομη είναι η διατύπωση ερώτησης, τόσο περισσότερο χρόνο έχει αρμόδιος ο Επίτροπος για να δώσει μια πλήρη απάντηση. Στον δεύτερο γύρο μπορεί να επιτραπεί μια συμπληρωματική ερώτηση εάν παραμένει τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την πρώτη ερώτηση και απάντηση. Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ο κάθε ομιλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει λοιπόν τη δική τους γλώσσα και φυσικά και ο υποψήφιος κ. Επίτροπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει διερμηνία, μην μιλάτε πολύ γρήγορα, ώστε να έχετε πλήρη διερμηνία των λόγων σας. Η συνολική ε, ακρόαση βρίσκεται στο διαδίκτυο στην, ε, σε web streaming και θα εμφανιστεί αργότερα και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και στο Twitter, στο hashtag EPHearings2014 μπορείτε να παρακολουθήσετε τα τεκτενόμενα. Και τώρα μετά από αυτές τις διευκρινήσεις θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαροσεύκοβιτς, τον υποψήφιο επίτροπο, για 15 λεπτά το maximum να κάνει τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις προς την Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας κύριε ε, Σεύκοβιτς και για τις δηλώσεις σας για το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρώπη, ώστε να υπάρξει πραγματικά προστασία της κινητικότητας αλλά και του κλίματος. Έχετε το λόγο.